Allora iniziamo le dichiarazioni di voto cominciando Εξηγήσεις ψήφου. Ξεκινάμε με την έκθεση του κυρίου Ριβελίνη για την απαλλαγή για το 2009 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο κύριος Ανάν. Thank you, madam. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ένα δί από εδώ, ένα δις από εκεί και σε λίγο θα αρχίσουμε να μιλάμε και για σοβαρά λεφτά. Τα λεφτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ε, διασώσεις οχριούν μπροστά στα έξοδα των ε, κυβερνήσεων μας. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε 7 δισεκατομμύρια στην Ελλανδία και τώρα θα δώσει άλλα 4,2 στην Πορτογαλία. Μιλάμε για παραπάνω από όλες τις εγχώριες περικοπές που κάναμε σε περικοπή του κοινωνικού κράτους. Και όλα αυτά για μια πολιτική η οποία προφανώ αποτυγχάνει. Όταν συμφωνήσαμε στην ελληνική διάσωση μα είπαν πω τώρα αποθαρρύναμε του κερδοσκόπου και η Ελλάδα θα μπορούσε να δανειστεί ανταγωνιστικά και δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Και βλέπετε πω η Ελλάδα ανοιχτά διαπραγματεύεται τη χρεοκοπία τη και περαιτέρω δάνεια. Είναι σαφέ πω δεν θα τα ξαναδούμε τα λεφτά μα αυτά και πως παραβιάζουμε τον νόμο. Οι διασώσει αυτέ δεν, όχι μόνο δεν εξουσιοδοτούνται από τη συνθήκη, απαγορεύονται ρητό. και είναι εκβιασμός των χωρών που δανείζονται, καθώς τράπεζες και κυβερνήσεις ε, κάνουν μια συμπεγνία για να δανείσουν τους ευρωπαϊκούς τραπεζίτες. Η Ελλάδα και η Ιρλανδία δανείζονται περισσότερα λεφτά για να στείλουν στην Πορτογαλία και αντιστρόφως. Και να τελειώσω να σας πω αυτό το οποίο είχε πει ο Ράντιαρτ Κίπλινγκ. Και η καλύτερη πολιτική είχε πει πως είναι να μην πληρώνουμε σε κανέναν για εκβιασμό, γιατί όποιο έθνος παίζει αυτό το παιχνίδι μόνο χάνει. Ευχαριστώ ο Φόξ. Uh, Κυρία Πρόεδρε, σήμερα ψηφίσαμε για, την, uh, για τους λογαριασμούς για τον προπολογισμό του 2009 και ψηφίσαμε μια εποχή όπου σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις πρέπει είναι αναγκασμένες να ε, υιοθετήσουν μέτρα λιτότητας, ε, μειώνονται οι μισθοί, αυξάνονται οι φόροι. Παράλληλα όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Επιτροπή ζητάει κάθε χρόνο και περισσότερα χρήματα. Και κάθε φορά το ελεκτικό συνέδριο αποφασίζει και λέει ε, ότι τα χρήματα αυτά δεν ξοδεύονται με τον σωστό τρόπο. Το ελεκτικό συνέδριο είπε ότι οι λογαριασμοί για το 2009 παρουσιάζουν πολλά λάθη. Γι' αυτό χαίρομαι που οι Βρετανοί συντηρητικοί και οι πολύ καλοί μας φίλοι Ευρωπαίοι συντηρητικοί καταψήφιζαν την απαλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίζει πολύ, με πολύ πιο προσεκτικό τρόπο τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ευχαριστώ κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όταν οι ψηφοφόροι μου με ρώτησαν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ένα από τα πράγματα που δεν καταλαβαίνουν, ειδικά σε καιρούς δύσκολους που περνάμε, είναι το γιατί ξοδεύουμε όλα αυτά τα λεφτά. Γιατί σε καιρό που οι κυβερνήσεις μας, η κυβέρνησή μας κάνει περικοπές, μειώνει τις δημόσιες δαπάνες και οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ένωση κάνουν ακριβώς το ίδιο, γιατί πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει περισσότερα λεφτά για τον προπολογισμό της, για τις μουσιονομικές προοπτικές και δεύτερον, γιατί δεν μπορεί να ξοδέψει τα λεφτά που έχει αποτελεσματικά. Όπως είπε και ο κύριος Φόξ, οι λογαριασμοί του 2009 είχαν πάρα πολλά λάθη. Δεν έχουν εγκριθεί εδώ και 15 και προσχώς 16 χρόνια. Και μας ρωτάνε οι ψηφοφόροι μας γιατί δεν ξοδεύουμε τα λεφτά τους καλύτερα πρέπει να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας. Ό,τι και να θεωρεί κανείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπωσδήποτε σωστό είναι να ξοδεύουμε με σωστό τρόπο τα λεφτά των προλογουμένων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάτεν είναι στην αίθουσα. Όχι. Δεν τον βλέπουμε, τον κύριο Μπάτεν, άρα περνάμε στην έκθεση Ήταλα για την απαλλαγή 2009 που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Τάκουλα έχει το λόγο. Parola all'onorevole Golni. O Kyrios Golnis. Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα την απαλλαγή για, αυτό του, για του Κοινοβουλίου, όχι για οικονομικού λόγου, αλλά για πολιτικού, διότι αυτό το Κοινοβούλιο είναι τα πάντα του από ένα Κοινοβούλιο. Δεν μιλάμε, δεν έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε, ακόμα και όταν τα θεμελιώδη δικαιώματα ενό μέλου του Κοινοβουλίου αμφισβητούνται. Πέραν του ατόμου μου, ε, ε, ντρέπομαι για το, για το Κοινοβούλιο, για το θεσμό μα αυτό. Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση ιδεών δεν υπάρχει καμία πραγματική ελευθερία έκφρασης. Είναι κομφορμισμό απλώς και μόνο. Κάνουμε μια δουλειά την οποία θα κάνανε πολύ καλύτερα μια τεχνική υπηρεσία εναρμόνιση ε, των προδιαγραφών και των κανόνων. Και κατά τα λοιπά παίζουμε σαν και μιμούμαστε την οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, ε, υπερασπίζουμε τα δικαιώματα στη Γουατεμάλα, στην Ινδονησία, εκεί όπου δεν έχουμε ε, κανένα δικαίωμα και καμία αρμοδιότητα, ενώ στη χώρα στην, στον τόπο μας δεν κάνουμε τίποτα. Ντρέπομαι πραγματικά για το Κοινοβούλιο διότι είναι αξιοθρύνητο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάκουλα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να φροντίσουμε να υπάρχει διαφάνεια και ε, προβολή του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να περικόψουν τους προπολογισμούς τους αυτή την εποχή και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει η διαφάνεια και το ανοιχτό πνεύμα σε όλα όσα κάνουμε. σε ό,τι αφορά τις περικοπές. Οι διάφορες καλλιτεχνικές υπηρεσίες, το βραβείο Λούξ, ουσιαστικά έχουν να κάνουν με κάποιες ε, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Και καλά κάνουν και υπάρχουν οι πόροι αυτοί, γιατί οι τέχνες, ε, ο πολιτισμός ε, είναι παραγωγή, για νεσιουργή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θα έπρεπε καλύτερα να περικόψουμε είναι η γραφειοκρατία και όχι η τέχνης και ο πολιτισμός. Θέλω να πω ότι Η μεταρρύθμιση των μισθών των βουλευτών ε, γίνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι ουσιαστικά, ο στόχος μάλλον, ε, μάλλον είναι, όλοι οι βουλευτές να έχουν λίγο πολύ τον ίδιο μισθό. Και το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και με τις φορολογικές τους πολιτικές στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Περνάμε στην έκθεση Μορέιρα για τις ε, αυτόνομες ε, εμπορικές ε, συναλλαγές για το Πακιστάν. Ο κύριος Ρόντε. Øh, Ευχαριστώ πολύ. Επισκεφθήκαμε, μάλλον όταν ψηφίσαμε την απόφαση για το Πακιστάν. Πρέπει κάποιος τώρα να χαίρεται που επιτέλους ψηφίστηκε αυτή η απόφαση. Είναι δύσκολη κατάσταση. Δήλθε μια πολύ δύσκολη περίοδο η χώρα αυτή. 415 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια έχει χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα και είναι πολύ καλό που αναλαμβάνουμε αυτή την πρωτοβουλία και έρουμε τους δασμούς από κάποια σημαντικά αγαθά όπως είναι τα κλωστοφαντουργικά προϊόντα και το, και το δέρμα γιατί ε, είναι μεν θετικό αυτό, αλλά είναι υποκριτικό και ατυχές να λέμε ότι αν σταματήσει αυτή η απαλλαγή ε, και ξαναβάλουμε τους ε, φραγμούς αυτούς, ε, θα έχουμε πρόβλημα. Ίσως είναι καλύτερο να καθυστερήσει η εφαρμογή της απαλλαγής. Ευχαριστώ κυρία Μοργάντη. Κύριε, συγγνώμη η ψηφοφορία αναβλήθηκε αλλά είμαστε αντίθετα, αντίθετοι με την έκθεση διότι δεν θέλουμε να ε, κλείσει ένας ολόκληρος βιομηχανικός τομέας ε, που είναι η κλωστοϊφαντουργία που ανέκαθεν ήταν η βάση των ε, βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Τοσκάνη. Τώρα μιλάμε για το Πακιστάν, αύριο μπορεί να μιλάμε για την Ινδία, για οποιοδήποτε άλλο κράτος. Αυτό είναι καρπός της επιταχυμένης εμπορικής πολιτικής του Πακιστάν. Μετά τις πλημμύρες ε, δώσαμε βοήθεια στο μισό εκατομμύριο στο, στο Πακιστάν και δώσαμε και μία ενίσχυση και για, ε, για, να, για να εμποδίσουμε τις δημοκρατικές παρεκκλήσεις ενδεχόμενα του Πακιστάν. Ε, μιλάμε για, και για τρομοκρατία, αλλά ε, μην ξεχνάμε και την δική, τις δικές μας ε, περιοχές. Το Βένετο πέρυσι πλημμύρισε και πολλές βιομηχανίες κλείσανε. Γι' αυτό θα θέλαμε να καταβληθούν προσπάθειες έτσι ώστε να έχουμε ε, δικά μας, δικές, δική μας παραγωγή. Η μικρή κλωστοϊφαντουργία οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί από την Ευρώπη στη μοίρα τους. Εκεί που παραγγείλουν, παραγγέλνουν μάλλον η ε, μεγάλη παραγωγή που έχουν μεταφέρει τα εργοστάσια τους αλλού. Εμείς όμως στη Λέγκα θέλουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας. Θέλουμε να σώσουμε τη γη μα. Μάρφη. Κύριος Μάρφη. Έξι μήνες μετά τις πλημμύρες στο Πακιστάν, ο ΙΕ μίλησε για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων. Πέρασαν άλλοι τρεις μήνες και είναι τελείως ανεπαρκής η απάντηση του ΠΟΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ υπερψήφισα του να δώσουμε επίγουσες ε, εμπορικές ε, προτιμήσεις ε, στο Πακιστάν, έτσι ώστε να μην είναι μόνο κάτι το συμβολικό που θα γεμίσουν τις ε, τσέπες ε, των κυβερνώντων. Ζητάω να δώσουμε αυτά τα λεφτά μέσω δημοκρατικών συνδικάτων για να πάνε στις περιοχές της πληγής Κάτι το σημαντικό μου επεσήμανε η Προοδευτική Ένωση Εργαζομένων του Πακιστάν. Είμαι κατά της απειλής της κυβέρνησης να μην επιτρέπει πλέον τον συνδικαλισμό σε εθνικό επίπεδο στο Πακιστάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η κυρία Μουσκαρντίνη δεν είναι στην αίθουσα, άρα περνάμε στην έκθεση Σούλτερ για τις μεταβατικές διατάξεις, για τις διμερείς συμφωνίες που επισυνάπτονται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τα τρίτα κράτη. Ο κύριος Αντωνιώτσι έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει άμεσες, ξένες ε, άμεσες επενδύσεις ε, στις δυνατότητες που προσφέρονται και, στην, ε, και η, σύμφωνα με την συνθήκη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα. Τώρα, επίσης σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, τα κράτη-μέλη ε, διατήρησαν ενισχύ τι διμερείς συμφωνίε που είχαν με τα τρίτα κράτη. Εάν δεν θέλουμε οι συμφωνίες αυτές να έρθουν σε αντίθεση με, την, ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας, δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε τις προτάσεις ε, του κ. Σούλτερ. Ε, ε, ή αυτά τα οποία προτείνονται ε, μας διασφαλίζουν, έναν, διασφαλίζουν μάλλον τους επενδυτές, προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και το σχέδιο αυτό κανονικά θεωρούμε ότι προχωρεί προς τη σωστή κατεύθυνση, γι' αυτό και το υπερψήφισα. Κύριε Σαντινόρο, Κύριε, κύριε Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή διότι είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι πρέπει να ελέγχουμε τι ευρωπαϊκέ επενδύσει στο εξωτερικό. Τώρα περνάμε κυρίω και αυδίω αυτή τη συγκυρία τη ε, οικονομική αστάθεια και ανασφάλεια. Τώρα θα πρέπει να δούμε ποιο έχει την αρμοδιότητα ε, για την προστασία από τι ποιε επενδύσει. Η ευθύνη ε, περνάει από τι εθνικέ κυβερνήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει προχωρήσει, ποιες είναι οι στρατηγικές γραμμές που θα ακολουθήσει. Πρέπει να προχωρήσουμε και με βάση την έγκριση των διμερών ε, ε, συμφωνιών και την διατήρηση της ισχύη των διμερών συμφωνιών θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να διαπραγματευτούν κάποιε ε, συμφωνίες και η Κομισιο... και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, επιβλέπει αν θέλετε την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων αυτών. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και μία κλιμάκωση αν θέλετε για το τι θα γίνει για τις συμφωνίες που έχουν ήδη ε, συναυθεί και τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει. Θα πρέπει επομένως να μην υπάρχουν νομικά, κοινά, ε, νομικά κενά και νομικές ασάφειες. Ε, ε, ε, εύχομαι για άλλη μια φορά η Κομισιό να μας κοινοποιήσει στο άμεσο μέλλον την στρατηγική που πρόκειται να ακολουθήσει έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν αυτά τα κενά. Λοιπόν, επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση του συναδέλφου Μορέιρα για την μακροοικονομική ενίσχυση της Γεωργίας. Κύριος Ρόντε. Vi har stemt om euro τα 46 εκατομμύρια που πρέπει να σταλούν στη Γεωργία ως ε, μακροοικονομική βοήθεια ε, συνοδεύονται με προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική ευθύνη και διαφάνεια. Αυτό είναι σημαντικό. Εξίσου σημαντικό είναι να έχουμε κατά νου ότι η πόρη αυτή, η κατανομή αυτών των πόρων είναι σημαντική και για μας γιατί έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία η Γεωργία μια χώρα η οποία επλήγει πρώτα απ' όλα από το πόλεμο με τη Ρωσία τον Αύγουστο του 2008 αλλά και από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση υπάρχει μάλιστα και εμπορικό εμπάργκο σε βάρος της από τη Ρωσία. Άρα είναι προς το δόφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει μια κυβέρνηση φιλική προ τη Δύση και μια κυβέρνηση που εφαρμόσει μεταρρυθμίσει. Αυτό κάναμε σήμερα. Ευχαριστώ. Η έχει λόγο. κύριος Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γεωργία είναι μια χώρα στρατηγικής σημασίας, ειδικά για τις ε, χώρες στο Ανατολικό και Νότιο μέρος της Ένωσης και επιπλέον καλύπτεται από την σχέση Ανατολικής Γειτονίας και είναι μια χώρα η οποία ακολουθεί μια ευρωατλαντική πολιτική σύγκρουση του 2008 έδειξε πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε η χώρα αυτή να μείνει εντό της ευρωπαϊκής σφαίρας. Το μακροοικονομικό σύστημα αυτό ενίσχυση, το οποίο εφαρμόστηκε από το 2009 παραμένει ένα στοιχείο κλειδί για την διεθνή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα της χώρας, οπότε συμφωνώ πλήρως με την απόφαση την οποία έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω κονδύλια προς την Γεωργία. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ πέρα η συζήτηση. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3 η ώρα.